Κατάξη 74, τρεις νομοθετικές πράξεις παραλαμβάνω και τώρα ε, έχουμε στη δυνάμει του 206 κάποιο διορθωτικό ε, από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και ε, λέει αυτή η διόρθωση ότι ε, σε σχέση με τη θέση του Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2011 όσον αφορά την θέσπιση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό όσον αφορά την ε, επιχειρησιακή διαχείριση κάποιων ε, ε, συστημάτων πληροφορικής σε μεγάλο ελληνικού στον τομέα ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε πρόκειται για κάτι πάρα πολύ πολύπλοκο όπως δείχνει και το όνομα αυτού του νομοθετήματος. Επίσης, Σύμφωνα με την διάταξη 22-16 4 αυτού διορθωτικού θα θεωρείται ότι εγκρίνεται 48 ώρε μετά την ανακοίνωση αυτή εκτό εάν υπάρχει κάποια ένσταση από πολιτική ομάδα ή από 40 συναδέλφου. Και θα γίνει η ψήφιση επίση ε, στο website του Κοινοβουλίου στο Σιάν Σαντιρέ.